της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας. Το λόγο έχει πάρει η κυρία Τίσον, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που μπορώ να ανακοινώσω την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ε, σχετικών με την προσβασιμότητα αποφάσεων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημαντική σας συμβολή, για τη σημαντική σας στήριξη καθ' όλη τη διάρκεια προετοιμασίας αυτής της πράξης. Ξέρετε πως ακόμα είναι πολλά τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν τα άτομα με αναπηρίες από την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων του στην κοινωνία. Πολύ συχνά δεν μπορούν να επιλέξουν ούτε πού ούτε πώς θα ζήσουν. Αντιμετωπίζουν επιπλέον προκλήσεις για να βρουν και να διατηρήσουν μια θέση εργασίας ή για να συμμετέχουν στην εκπαίδευση για να απαραθέσουν μόνο μερικές από τις δυσκολίες. Η τεχνολογική καινοτομία προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια. Έχουμε το ηλεκτρονικέ τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, τα έξυπνα τηλέφωνα, τα smartphone δηλαδή. Αλλάζει η κοινωνία μας και γίνεται η ζωή μας πιο εύκολη. Αυτά τα προϊόντα και αυτές οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες και προσφέρουν νέες ευκαιρίες σε άτομα τα οποία έχουν αναπηρίες για να συμμετέχουν στην κοινωνία και για να ζουν ανεξάρτητα. Βλέπουμε πως η ζήτηση για τέτοιου είδους προσβάσιμα προϊόντα αυξάνεται και αυτό εντείνεται και από την γύρανση του πληθυσμού. Μέχρι το 2020, 120 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα έχουν περιορισμούς λειτουργικούς ή αναπηρίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει τη δέσμευση και αυτό έγινε μέσω των συμβάσεων του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίες να κατασκευάζουν προϊόντα, να ετοιμάζουν υπηρεσίες και κτίρια τα οποία θα είναι πιο προσβάσιμα. Τα κράτη-μέλη έχουν ξεκινήσει να νομοθετούν για το θέμα αυτό της προσβασιμότητας ανεξάρτητα και χωρίς συντονισμό. Αν λοιπόν δεν δράσουμε εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι διαφορές ε, στα εθνικά δίκαια κάθε κράτους μέλους θα αυξηθούν με αποτέλεσμα για τη βιομηχανία να γίνει όλο και πιο δύσκολο να πόλουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίε τους εκτός των συνόρων τους και βεβαίως θα είναι όλο και λιγότερες οι σε όλη την Ευρώπη προσβάσιμες υπηρεσίες και τα προσβάσιμα προϊόντα. Έχουμε λοιπόν ως στόχο να περιορίσουμε και να προλάβουμε τα εμπόδια μεταξύ κρατών μελών που θα δημιουργούσε αυτή αυτές οι διαφοροποιημένες και διαφορετικές απαιτήσει των εθνικών νομοθεσιών. Θέλουμε λοιπόν λειτουργικότητα και προσβασιμότητα βασιζόμενη σε ένα κοινό σχεδιασμό που θα επιτρέψει στη βιομηχανία μας να προτείνουν μια μεγαλύτερη γκάμα προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών σε καλύτερες τιμές σε όλη την Ευρώπη. Οι λειτουργικές απαιτήσεις που έχουμε συμπεριλάβει στο, στην πράξη αυτή βασίζονται σε κάποιες αρχές προσβασιμότητας και δεν περιγράφουν με λεπτομέρεια τις τεχνικές λύσεις που θα επιλεγούν. Αυτό αφήνει περιθώριο στην καινοτομία και μπορούμε με τον τρόπο αυτό να είμαστε και πιο ευέλικτοι. Μετά από πολύ εντατικέ διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενου και τους ενδιαφερούμενου φορείς έχουμε επιλέξει κάποια προϊόντα κλειδιά, κάποιε κομβικές υπηρεσίες από την καθημερινότητα που είναι τα πιο σχετικά και που χρειάζονται περισσότερο για να στηρίξουν την ανεξάρτητη διαβίωση. Και α είμαστε ειλικρινεί. Όλοι όλων η ποιότητα ζωή μπορεί να βελτιωθεί από μικρές βελτιώσεις στο επίπεδο προσβασιμότητας που έχουμε. Για παράδειγμα, θα είναι καλύτερο για εμάς να ακούμε καλύτερα τις ανακοινώσεις του σταθμού των τρένων είναι προτιμότερο το μεγάλο φορμάτ που θα μας επιτρέπει πιο εύκολα να διαβάζουμε ανακοινώσεις. Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις και κυρίως τις μικρομεσαίες να προωθούν σε άλλα κράτη-μέλη τα προϊόντα τους. Έτσι θα ενθαρρύνουμε το διασυνοριακό εμπόδιο και θα βελτιώσουμε τον ανταγωνισμό. Θα πρέπει οι δημόσιες αρχές όταν προετοιμάζουν διαγωνισμούς για υπηρεσίες κτίρια ή προϊόντα να γνωρίζουν ποιες είναι οι απαιτήσει τις οποίες θα πρέπει να σεβαστούν κατά την προσφερά τους εταιρείε. Έχουμε επίσης και μία ρήτρα κοινή σε αυτές τις διατάξεις που θα εξασφαλίσουν την αναλογικότητα, την ισορροπία, θα προωθήσουν τις ε, πολύ μικρές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα λάβει όλες τις δέσους ε, διατάξεις υπόψη. Έχουμε το σχέδιο οδηγίας για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων των δημοσίων φορέων, για τον οποίο έχετε ήδη γνωμοδοτήσει. Προχωράει και η οδηγία προσβασιμότητα στο Συμβούλιο έχει φτάσει στο επίπεδο όπου ελπίζουμε πως ο τριμερής διάλογος σε λίγο θα ξεκινήσει. Ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει με την επικοδομητική και θετική προσέγγιση που έχει επιλέξει και να μας βοηθήσει να εγκρίνουμε την ομοθεσία το συντομότερο δυνατόν. Πιστεύω πως εδώ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που μας ευνοεί όλους. Είναι win-win και χάρη στην πρόταση αυτή το κόστος για τα κράτη-μέλη και τις επιχειρήσεις θα μειωθεί και επιπλέον η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επηρεάσει θετικά και τους δημόσιους προϋπολογισμούς μακροπρόθεσμα, μειώνοντας την εξάρτηση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία. Και το πιο σημαντικό είναι η οδηγία αυτή θα διευκολύνει την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες στην παιδεία, θα τους δώσει περισσότερες εργασιακές ευκαιρίες, θα τους προσφέρει περισσότερη ελευθερία, πιο πολλές ευκαιρίες στην καθημερινότητά τους. Θα κλείσω τονίζοντας για μία ακόμα φορά πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάθε πρόθεση να ενισχύσει την κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Κανείς δεν θα πρέπει να μείνει πίσω. Η πρόταση αυτή τονίζει την υποχρέωση και τη δέσμευση που έχουμε να αναλάβει η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική πρόοδος να συνοδεύουν η μία την άλλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Από το ΕΛΚ η κυρία Εστερά Φαραγκούτ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την Επίτροπο την κυρία Τίσεν. Η οδηγία αυτή πραγματικά είναι πολύ δημοφιλής και εγώ έλαβα πάρα πολλές ερωτήσεις για το πότε θα εγκριθεί. Από το 2012 την περιμένουμε. Συγχαρητήρια λοιπόν προσβασιμότητα είναι η λέξη κλειδί για όλα και κυρίως για την κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρίες, γιατί είναι μια προϋπόθεση για να μπορούν με ισότιμο τρόπο να συμμετέχουν πλήρως ε, στην κοινωνική ζωή των ατόμων με περιορισμένη λειτουργικότητα. Είμαστε μια μεγάλη αγορά που θα πρέπει να έχει προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίε, μειώνοντα τα εμπόδια που έχει δημιουργήσει η ισχύουσα νομοθεσία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κατάτμιση νομοθετική και κανονιστική και κάθε κρατός μέλος αυτή τη στιγμή ρυθμίζει μόνο του τα θέματα αυτά. Έχουμε τη σύμβαση του ΟΗΕ που στα τελικά συμπεράσματα μίλησε για την εφαρμογή της σύμβασης για άτομα με αναπηρίες στο εδάφιο 9 που θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα. Έχουμε τραπεζικές υπηρεσίες, τηλέφωνα, υπολογιστές, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. Είναι μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών και νομίζω πως η παρατήρηση 29 των Ηνωμένων Εθνών για το φυσικό περιβάλλον, για την επικοινωνία και για το σχεδιασμό θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη. Ευχαριστώ κυρία Γιούτα Στάινρουκ. κανένα λεπτό, Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Η πρόταση της Επιτροπής για την βελτίωση της ε, ε, προσβασιμότητας σε παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες είναι πάρα πολύ σημαντική για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη. Βεβαίως και υπάρχουν κοινέ προδιαγραφές και κοινή αντιμετώπιση απλουστευμένη ε, πρόσβαση λοιπόν και εξοικονόμηση από τις δαπάνες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή η βελτίωση της προσβασιμότητας προβλέπεται άλλωστε στο, Σύμφωνο, των Ομένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που προβλέπει την ε, ισότιμη πρόσβαση ε, στον ίδιο βαθμό με την ενεργό ενσωμάτωση στις κοινωνίες. Το ίδιο νομίζω πρέπει να ισχύει για κάθε τομέα της ζωής, ώστε να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να ενσωματώνονται και στην αγορά εργασία το ταχύτερο και καλύτερο δυνατό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μάκιντάιρ, ECR, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα την ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο να υποδεχθώ μεταξύ άλλων τον Κάλεμ Ράσελ που ήρθε σε μια εκδήλωσή μας να μιλήσει για τις ευκαιρίες για νέους με αναπηρία. Ο Κάλεμ είναι φοιτητή στο Κολέγιο της Ευρώπης της Βρύγης. Ένας νέος, αποφασισμένος, ταλαντούχος, βρετανός, τυφλός. Η αναπηρία όμως δεν μπορεί να προσδιορίζει έναν άνθρωπο. Η αναπηρία δεν μπορεί να αποτελεί φραγμό στο να διαδραματίζει κανείς πλήρη ρόλο στην κοινωνία. Ο Κάλεμ λοιπόν επισήμανε ότι οι ιστοσελίδες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως απροσπέλαστες για άτομα με αναπηρίες. Για όνομα του Θεού λοιπόν ας αντιμετωπίσουμε πρώτα τα δικά μας, τα του δικού μας οίκου. Όπως λέμε και στα αγγλικά, όποιος ζει σε γυάλινο σπίτι ας μην πετάει πέτρες. Ας αρχίσουμε λοιπόν από την προσβασιμότητα των δικών μας ιστοσελίδων και ιστοτόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά ας πούμε παραπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χάρκιν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ και καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ κυρία Επίτροπε γιατί κάνατε αυτό που είπατε ακριβώς. Δηλαδή ε, έχετε εισαγάγει μία ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας, έτσι ώστε όσοι έχουν αναπηρίες να έχουν καλύτερη προσβασιμότητα. Θα έχουμε 120 εκατομμύρια ανθρώπους μέχρι το 2020 με κάποια μορφή αναπηρίας. Γι' αυτό θα κάνουμε πολύ καλό στους ανθρώπους με αναπηρία, αλλά έχει και νόημα οικονομικά. Δηλαδή θα έχουμε περισσότερους ε, πελάτες στις επιχειρήσεις μας. Μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, τραπεζικές υπηρεσίες, e-books, smartphones, ε, τηλεοράσεις και υπηρεσίες μεταφορών. Τα πάντα περιλαμβάνονται. Και όπως είπατε και εσείς, ε, θα πρέπει να βρεθούν τεχνικές λύσεις που δεν είναι λεπτομερείς. Εδώ μιλάμε για τα γενικά χαρακτηριστικά που διέπουν τις υπηρεσίες και τα αγαθά τα οποία ορίζονται σωστά. Νομίζω ότι θα πρέπει να ορίσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά για τους κατασκευαστές και τις επιχειρήσεις. Έχουμε επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων ε, Εθνών για τους ανθρώπους με αναπηρίες και αυτό αποτελεί προ κρίμα. Γινόμαστε μια ψηφιακή κοινωνία και έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και για τον μη αποκλεισμό στον ψηφιακό τομέα. Για την ΓΚΟΕ, η κυρία Μαρτίνα Άντερσον για ένα λεπτό. Αφού ασχολήθηκα στο Ντέρι με θέματα αναπηρίας και μετά από την έρευνα των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με την παραβίαση των δικαιωμάτων ανθρώπων ε, με αναπηρία, βλέπουμε ότι γίνονται περικοπές και στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι περικοπές έχουν ε, πλήξει περισσότερους ανθρώπους με αναπηρία. Τι γίνεται με τα 80 εκατομμύρια αναπήρους που πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ATM, στις μεταφορές, στις τραπεζικές υπηρεσίες, τους υπολογιστές. οι βουλευτές χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες για να έρθουν εδώ στο Στρασβούργο. Εγώ τις χρησιμοποιώ. Μια πράξη προσβασιμότητα θα επέβαλε στα κράτη-μέλη να νομοθετήσουν για τα άτομα με αναπηρία μέσα στα πλαίσια και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών που η Ιρλανδία θα πρέπει να κυρώσει. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Από τη δική μου ομάδα των Πρασίνων δεν είναι ο μιλητής ε, στην αίθουσα, ο κύριος Στάρλαντ δηλαδή, και άρα δίνω το λόγο στον κύριο Κώσα για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί κρατήσατε την υπόσχεσή σας και σε λιγότερο από ένα χρόνο προβάλατε και συντάξατε αυτή την πράξη προσβασιμότητας. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε για τα προσκόμματα που υπάρχουν. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι προσβάσιμη. Τονίσατε το ότι μέχρι το 2020 θα έχουμε 120 εκατομμύρια ανθρώπους με κάποιο είδος αναπηρίας. Δηλαδή ένας στους τέσσερις πολίτες της Ευρώπης θα έχει κάποιο είδους αναπηρία ο κανονισμός για τα ευρωπαϊκά ε, ταμεία είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτού του φάσματος ή του πακέτου, καθώς και ο χάρτης για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες, ιδιαίτερα η σύσταση παριθμών 2. Θα ήθελα να πω ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε στο ευρωπαϊκό δίκαιο έναν ορισμό σε σχέση με την προσβασιμότητα. Και αυτό αποτελεί ένα πλαίσιο για την εργασία μας. Είναι μακρύς ο δρόμος, πρώτα θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ, αλλά μετά από πέντε χρόνια μπορούμε να αρχίσουμε την ε, πραγματική εργασία. Τέλος, ε, εν κατακλείδη, θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να καλωσορίσω το γεγονός ότι θα έρθουν όλα αυτά τα προσκόμματα. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Κάθριν Στήλερ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επίτροπο. Καλωσορίσω λοιπόν την πρόταση για την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας που όπως είπαν ε, πολλοί έκανε μακρύ δρόμο μέχρι να φτάσει εδώ αλλά είναι πολύ σημαντική λαμβάνοντα υπόψη ότι χρειάζεται ε, να έχουν ε, πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες οι συμπολίτε μας με αναπηρία που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα λοιπόν θέλω να καλωσορίσω τα θέματα που αφορούν το, τα λειτουργικά συστήματα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές γενικότερα, αλλά βέβαια και τη λειτουργικότητα των, ιστοσε, ιστοτόπων που ανέφερε και η Επιτροπός και βέβαια το θέμα των ιστοτόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς από την Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς φροντίσαμε τουλάχιστον οι δικές μας ιστοσελίδες να είναι προσβάσιμες και κάνουμε ό,τι μπορούμε πάντα. Οι προτάσεις αυτές λοιπόν που θα εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει διάκριση και στην ψηφιακή εσωτερική αγορά είναι πολύ σημαντικές για όλους τους πολίτες. Τα Ηνωμένα Έθνη προτείνουν την ε, αναθεώρηση από δεκαετία των προτάσεων για την κοινωνία της πληροφορίας και υπογραμμίσουν 12 συγκεκριμένα προβλήματα ή προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε σχέση με την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τόσο εμείς λοιπόν όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα σε τα θέματα αυτά. Η συνθήκη του Μαρακές καλύπτει τα ζητήματα αυτά και καλό την Επιτροπή να υιοθετήσει νομοθετική πρόταση για την υλοποίηση αυτής της συνθήκης του Μαρακές ε, ιδιαίτερα το θέμα των ηλεκτρονικών βιβλίων, e-books, που είναι ε, που ε, σε πολύ περιορισμένο βαθμό μόνο 5% δημοσιεύονται σε με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι προσβάσιμα για άτομα με τύφλωση ή με δυσκολίες όρασης, ενώ στις πιο φτωχές χώρες είναι μόλις 1%. Έχουμε λοιπόν αυτό το σημαντικό ορόσημο μπροστά μας, στην υλοποίηση συνθήκης του Σε Ευχαριστώ πολύ, Χέλγα Στίβενιτς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με την πρόταση αυτή για την προσβασιμότητα. Υπάρχει μόνο ένα κομμάτι αυτής που αναφέρεται στην σύμβαση του ΟΕΕ για άτομα με αναπηρίες. Ελπίζω λοιπόν πως θα κάνει ό,τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει τα πράγματα και σε άλλους κλάδους που χρειάζεται αυτό. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εσωτερική αγορά που να καλύπτει τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε σε όλα τα εμπόδια τα οποία ακόμα παραμένουν. Θα μιλήσω για τους ιστοτόπους όπου είναι αυξημένο το κόστος αν οι επιχειρήσεις θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους ε, σε όλη την Ευρώπη, καλύπτοντας τους εθνικούς κανόνες ε, σε κάθε περίπτωση. Ποια είναι τα συμφέροντα των καταναλωτών, ποια είναι τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, πώς μπορούμε να προωθήσουμε και να προκρίνουμε την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη των ατόμων με αναπηρίες, γιατί ξέρουμε πως θα αυξηθεί αυτό το τμήμα του πληθυσμού στα 120 εκατομμύρια μέχρι το 2020, γιατί ο πληθυσμός μας γυράσκει. Θέλουμε λοιπόν μια ευρωπαϊκή πράξη η οποία θα είναι ε, έτοιμη να επηρεάσει τη ζωή μας και τώρα. λεπτό η κυρία Σαράσοβα. Τα 80 εκατομμύρια πολιτών με αναπηρίες χρειάζονται και αξίζουν ίση πρόσβαση όχι μόνο στην ε, αγορά αλλά και στην ψηφιακή αγορά, για να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες. Χαίρομαι για την πράξη πρόσβασιμότητας, αλλά περιμένοντας για μακρό χρονικό διάστημα αυτή την πρόταση θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε σε έμπρακτα αποτελέσματα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις. Ε, αυτό θα πρέπει να γίνει πράξη για τους ανθρώπους στην καθημερινή του ζωή. Επειδή ασχολήθηκα με την οδηγία για την προσβασιμότητα του διαδικτύου, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια βρίσκεται, ποιος βρίσκεται ότι είναι ο συσχετισμός μεταξύ των δύο κειμένων. Νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερες διασαφηνίσεις πριν μπούμε στον τριμερή διάλογο το νέο έτος. Το Κοινοβούλιο δεν θα παρετηθεί ζητώντας καλύτερη και περισσότερη προσβασιμότητα σε σχέση με την κάλυψη και του διαδικτύου. Χρειάζεται πλήρης πρόσβαση στο διαδίκτυο και την εσωτερική αγορά. Δεν μιλάμε μόνο για τους δημόσιους ιστοτόπους. Φτάνουμε τώρα στο τελευταίο κάτω. Κάτσε της μας με την κυρία Σότροβα ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ένα πράγμα θέλω να πω. ότι θέλω να υποστηρίξω τα λόγια σας. στο τέλος της ομιλίας σας ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα άτομα με αναπηρία. Αποτελεί αυτή εκ των όνων προϋπόθεση για την πρόσβαση και στις λοιπές υπηρεσίες και την πλήρη αξιοποίηση τους φερειπίν ψηφιακές υπηρεσίες. Όλοι συμφωνούμε πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίζεται η προσβασιμότητα. Πάντως πρόβλημα προκύπτει όταν έρχεται η ώρα να αναστήσουμε πόρους. Ξέρουμε πολύ καλά και από τους εθνικού μας προπολογισμού. πόσο δύσκολο είναι αυτό. Πρέπει λοιπόν να προβάλλεται πάντα το επιχείρημα ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης και η πρόσβασιμότητα στην εκπαίδευση αυτή αποτελεί καθήκον και επένδυση. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό. Η επόμενη μιλήτρια. Κύριε Σεχνάλοβα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε. Η ευρωπαϊκή αυτή πράξη προσβασιμότητας είναι καλωρή, καλοδεχούμενη, παρόλο που αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και το είδαμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το είδαμε και κατά τη συζήτηση της ε, οδηγίας για τον Ευρωπαϊκό Ιστότοπο είναι ένα έγγραφο το οποίο δημιουργεί πάρα πολλές προσδοκίες για τα άτομα με αναπηρίες και ελπίζω πως αυτές δεν θα συνθλιβούν. 80 εκατομμύρια ατόμων με αναπηρίες αντιμετωπίζουν πάρα πολλά εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται αυτή η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που θα βελτιώσει τη ζωή τους, όπως και τη ζωή των ηλικιωμένων. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τους οποίους θα θέλαμε να στηρίξουμε αυτή την πράξη και ελπίζουμε πως τα κράτη-μέλη θα κάνουν το ίδιο. Ο κύριος Μαριάς είναι ο τελευταίος ομιλητής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάνω από 80 εκατομμύρια άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποια μορφή αναπηρίας θεωρούμε λοιπόν σημαντική την πρωτοβουλία για τη θέσπιση ευρωπαϊκής οδηγίας για την προσβασιμότητα των αναπήρων στην εκπαίδευση στο εμπόριο στην εργασία ενισχύοντας έτσι την κοινωνική δικαιοσύνη. με βάση τα στοιχεία της eurostat ένα άτομο σε παραγωγική ηλικία έχει πιθανότητα 66% να βρει δουλειά ενώ για ένα άτομο με βαριά αναπηρία η πιθανότητα μειώνεται στο. είκοσι στη χώρα μου την ελλάδα το ποσοστό ατόμων με αναπηρία ανέρχεται στο 10% του πληθυσμού ενώ σύμφωνα με την ελστάτ το 84% των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μου βρίσκονται εκτό αγορά εργασία. το μνημόνιο και οι πολιτικέ λιτότητας εξουθένωσαν ακόμη περισσότερο τα άτομα με αναπηρία καθώ βρέθηκαν στο στόχαστο τη τρόικα η οποία του μείωσε τα προνοιακά επιδόματα και τι αναπηρικές συντάξει, που πλέον κυμαίνονται από διακόσια πενήντα έως πεντακόσια ευρώ οδηγώντας έτσι τα άτομα με ειδικές ανάγκες στον κοινωνικό αποκλεισμό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα η κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Νιώθω σαν να είμαι συνάδελφος εδώ, μέλη λοιπόν του Κοινοβουλίου, ευρωβουλευτές, αγαπητοί ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας. Πραγματικά θέλω να συνεργαστούμε και ευελπιστώ ότι αυτό το πακέτο θα ολοκληρωθεί νωρίτερα από ό,τι περιμένουμε και θα εφαρμοστεί επίσης έγκαιρα θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσβασιμότητα για όλους τα μέσα που ε, διαθέτουμε. Και αυτό αφορά και τα ε, στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι όλα τα στοιχεία του πακέτου θα είναι προσβάσιμα σε ανθρώπους με αναπηρίες για να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη η Helga Stevens είπε ότι είναι πολύ καλή ε, πρόταση, αλλά σημαίνει πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν επίσης ε, συγκεκριμένα στοιχεία ως προς το κόστος, αλλά προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε αρκετά χαμηλό, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν επιλογές. Επίσης προσπαθήσαμε να φτάσουμε σε ένα σχεδιασμό για όλους ένα σχεδιασμό που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους. Λαμβάνουμε υπόψη νέες υπηρεσίες και νέα προϊόντα, άρα δεν μιλάμε για ε, αναθεωρήσει μεταρρυθμίσεις στοιχείων που ήδη υπάρχουν ή μεθόδων που υπάρχουν. Το κόστος προσπαθούμε να το συμπιέσουμε και αν είναι παρόλα αυτά υψηλό, θα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί το θέμα της προσβασιμότητας είναι πολύ σημαντικό. Εάν θα πρέπει να αλλάξει μορφή το αρχικό προϊόν, τότε η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε κάτι το διαφορετικό. Το προϊόν όμως θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές μας. Είδαμε το θέμα του κόστους για τη βιομηχανία, αλλά θα θέλαμε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να είναι προσβάσιμα σε όλους, να πληρούν τις προϋποθέσεις και αν το υποστηρίξουμε όλοι, ίσως θα υπάρχει χαμηλότερο κόστος, συμπιεσμένο κόστος και θα έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας ως προς τη, τις ε, λειτουργικές ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, καθώς και με την εμβέλεια της πράξης. Θα πρέπει να αρχίσει ο τριμερής διάλογος, έχουμε την οδηγία. Μιλάμε για ιδιωτικά, ιδιωτικούς ιστοτόπους και δημόσιους, αλλά το λειτουργικό θα είναι το ίδιο σε σχέση με τα ε, πνευματικά δικαιώματα. Η κυρία Στάιλερ το αναφέρε αυτό. Η συμφωνία του Μαρακές ε, προβλέπει μια εξαίρεση για τα τυπωμένα βιβλία. Εάν θέλετε να έχετε και μία έκδοση σε μπράι, εδώ μιλάμε για e-books και όχι τυπωμένα βιβλία, τα οποία μπορεί κανείς να κατεβάσει και θα θέλαμε να υπάρχει προσβασιμότητα για ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα υπάρχει προσβασιμότητα και για τους τυφλούς και για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Κάτι το οποίο έχουμε κάνει εξ αρχής. Θα υπάρχει ένα μικρό κόστος ε, προσαρμογής, αλλά θα υπάρχει καλύτερη προσβασιμότητα. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνεται έτσι